Τριμερή ημερήσια διάταξη τώρα και πρώτα απ' όλα έχουμε την έκθεση του κυρίου Σάιον για την εξουσία ανάθεση νομοθετικού έργου. Το λόγο έχει ο εισηγητή πρώτο. Εξότιμη Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτ, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή. πολλοί ξεκινούν τις παρεμβάσει τους εξηγώντα πόσο σημαντικό είναι το θέμα του ή υπογραμμίζοντα ότι είναι το πιο σημαντικό, τη καταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων. Επιτρέψτε μου όμω να πω ότι εγώ διεκδικώ πολύ πιο σοβαρούς λόγους για τη σημασία την οποία θα ήθελα να αναγνωρίσετε στο δικό μου θέμα έκθεσης. Ίσως είναι ένα από τα και πιο σημαντικά αλλά και πιο ε, σπάνια αν θέλετε χαρακτηριστικά της νέας αυτής συνθήκης της Λισαβόνας. Εκείνοι οι οποίοι είχαν επικρίνει ε, τις προτάσεις συνθήκης ε, της Λισαβόνας ε, είχαν αγνοήσει την πρόταση για το δικαίωμα αυτό, δηλαδή το δικαίωμα της εκχώρησης της ανάθεσης νομοθετικού έργου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ότι οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί απευθείας από τον πολίτη έχουν και την εντολή από τον πολίτη της Ευρώπης για την ε, παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής μέσω των κανονισμών ή των οδηγιών. Μπορούν δηλαδή να ελέγχουν την Επιτροπή στους κανονισμούς και τις οδηγίες που ε, εισάγει και ταυτόχρονα μπορούν και να την προλαβαίνουν. Αυτές είναι οι διαδικασίες που προτείνει, που προβλέπει μάλλον η διαδικασία τη συναπόφαση. Ταυτόχρονα, ναι, διευρύνονται το πεδίο αυτό των ε, αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα όμως η ποιότητα του νομοθετικού μας έργου δεν εξαρτάται μόνο από τη συναπόφαση από τα θέματα που θα υπάρχουν σε αυτήν, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσουμε το νομοθετικό μας καθήκον. Έχουμε λοιπόν σε αρκετά από τα νομοθετήματα που έχει εξετάσει το Κοινοβούλιο φτάσει σε ένα επίπεδο κατά το οποίο μπορούμε να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τις αποφάσεις για την περαιτέρω εκτέλεση των νομοθετημάτων αυτών υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό στο παρελθόν μέσα από μια διοργανική συμφωνία είχε επιληθεί μέσα από μια διαδικασία η οποία όμως δεν επέτρεπε ουσιαστικό έλεγχο της περαιτέρω ε, δράσης της Επιτροπής. Τώρα όμως μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και το άρθρο 92 αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων των βουλευτών. Διότι αν εμείς οι βουλευτές λαμβάνουμε σοβαρά, στα σοβαρά τα καθήκοντά μας και θέλουμε να ασκήσουμε πραγματικά την λειτουργία μας ε, ως οργάνου συναπόφασης και προσπαθώ να εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτή η διαδικασία, θα μπορούσαμε να καλύψουμε και το δημοκρατικό λεγόμενο έλλειμμα Το Συμβούλιο λοιπόν και το Κοινοβούλιο δεν μπορούν να ρυθμίσουν το κάθε παραμικρό ζήτημα που προτείνει από το νομοθεσία του. Το Κοινοβούλιο έχει ολομέλεια μια φορά το μήνα. Συνεδριάσει όπω η σημερινή μα δείχνουν ότι υπάρχουν και δυσκολίε πρακτικέ όπου δεν μπορούν όλοι να είναι και παρόντε. Πλην όμω μπορεί το Κοινοβούλιο να ελέγχει και να παρακολουθεί τα ζητήματα τα οποία έχει, για τα οποία έχει εκχωρήσει το νομοθετικό έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι δυνατόν πλέον με το η νέα συνθήκη και ταυτόχρονα διαφυλάτει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ελέγξει ότι πράγματι τηρούνται όλες οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συνθήκη και ότι μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ανα πάσα στιγμή. Αυτή είναι μια εγγύηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημοκρατικών διαδικασιών των ε, δημοκρατικών οργάνων και Βεβαίω χρειάζεται Συμβούλιο και Επιτροπή να κάνουν και τη δουλειά του από τη δική του την πλευρά, αλλά σημαντικό στην νέα κατάσταση είναι ότι διαφυλάτουν τα δικαιώματά του, μάλλον τι προνομίε του, τα αρμόδια για την ομοθεσία, όργανα, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει επίτροπο κ. Σεφσοβιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σάιτζεκ για την ιδιαίτερα αποτελεσματική έκθεση την οποία συνέταξε και να ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για το ζήτημα με το οποίο αντιμετωπίζει το θέμα των ε, πράξη, των πράξεων κατεξιοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε όλο αυτό το ζήτημα, αλλά χρειάζονται κάποιε κατευθυντικέ γραμμέ προκειμένου να ε, αποφύγουμε μια εξέταση μάλλον να εφαρμόσουμε μια εξέταση πιο αποτελεσματική. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια πιο πρακτική προσέγγιση στην ε, μελλοντική νομοθεσία. Θα ήθελα να γραμμίσω την ε, σημασία που αποδίδει η Κομισιόν στην ε, διοργανική συμφωνία σε θέματα πράξεων κατεξιοδότηση. Επί της θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Κομισιόν καλωσορίζει την έκθεση, μπορεί να διαφωνεί σε κάποια ζητήματα, αλλά βασικά έχουμε τον αυτό στόχο. Θέλουμε αποτελεσματικότητα, σαφήνεια, διαφάνεια και μια εξορρόπηση των αρμοδιοτήτων. Αν μου επιτρέπετε να καταστώ λίγο πιο συγκεκριμένο, θα ήθελα να κάνω κάποιε σύντομε παρατηρήσει σε ορισμένα σημεία. Σε ό,τι φορά τώρα τον ε, θέμα του άρθρου 290, ιδιαίτερα στην δεύτερη παράγραφο, εδώ έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τα μέσα ελέγχου του νομοθέτη σε θέματα ε, ε, των πράξεων αυτών. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποιες πρακτικές λύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διάρκεια της ε, εκχώρησης αρμοδιοτήτων θα θέλαμε εδώ να συμφωνήσουμε με την ε, σιωπηρή ε, έγκριση διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επαντηλημένα μας έχει βοηθήσει στην νομοθεσία τόσο τη διάρκεια το θέματος ε, της ένστασης και εδώ θα πρέπει να πω ότι συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή για τους δύο μήνες συν δύο επιπλέον μήνες ε, παράτασης. Ε, νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε και τα τρία θεσμικά όργανα. Και ήδη έχουμε κάποια παραδείγματα σχετικά με το πώς έχει ήδη εφαρμοστεί στο πλαίσιο της νομοθετικής δράσης. Τώρα, σε ό,τι φορά το θέμα του επίγοντος ή κατεπίγοντος, έχουμε κάποια παραδείγματα από την ιστορία σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη το ζήτημα τη ασφάλεια των τροφίμων, ασφάλεια των παιχνιδιών. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιε διαδικασίε και απαιτείται να βρούμε κάτι το πιο σαφέ από την πρόταση που κάνει ο εισηγητή. Για αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω σχετικά με το ζήτημα της ευθυγράμμιση να αναφερθώ εδώ στην πραγματιστική προσέγγιση, διότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν δούλεψαν σημαντικά σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση των 350 ε, νομοθετικών πράξεων που έχουν ευθυγραμμιστεί σύμφωνα με την προσέγγιση Πράγκ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει αυτή η προσέγγιση, κάτι η οποία δεν είχε επιτευχθεί μέχρι τώρα σύμφωνα με την αρχή της, ε, του ελέγχου του κανονιστικού ελέγχου, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα, εξ ονόμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, το λόγο έχει ο Πρόεδρος, κύριος Λάινεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίμενε εδώ και καιρό για να είμαστε ισότιμοι με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του ελέγχου ε, νομοθετημάτων που έχουμε χωρίσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να σας εξηγήσω λίγο, το έτος 2008 είχαμε 6.000 νομοθετήματα χωρίσει, δηλαδή βουνό ολόκληρο κανόνων που ε, σε ένα είδο δευτερεύουσα δευτερογενού νομοθεσία περνούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παλιά διαδικασία της Επιτροπολογίας και διεκπεραιωνόταν εκεί. Ε, εμείς είχαμε πολύ λίγα δικαιώματα, μας ενημέρωναν μεν, αλλά δεν ήμασταν συνομοθέτες. Και τώρα το κατάφερε επιτέλου η συνθήκη της Λισαβόνα. είμαστε επίσης με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ε, του ελέγχου ε, των ε, νομοθετημάτων που εκχωρούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλουμε ε, να είμαστε πλήρως ισότιμα μέλη. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Επιτροπέ, όταν λέτε να υπάρχει δυνατότητα του κατεπήγοντος, αλλά θα πρέπει εγκαίρως και πολύ γρήγορα να ενημερώμαστε ταυτόχρονα με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε τώρα στους ομιλητές εκπέρους των ομάδων. Ο πρώτος είναι ο κύριος Κοέλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, κατά την άποψή μου θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον στέλφο Σάιγερ για την έκθεσή του. Η συνθήκη Λισαβόνα ενισχύει τι εξουσίε του Κοινοβουλίου και πραγματικά αυξάνει τον ε, δημοκρατικό έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι διπλά ευγνώμων προς τον κύριο Σάγερ ε, για την έκθεση την οποία συνέταξε αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θέτουμε τέρμα στην παλιά επιτροπολογία που πολύ συχνά είχαμε επικρίνει στο Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε το άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας ε, και η έκθεση του συναδέλφου Σάγερ περιέχει διάφορες ε, προτάσεις διαδικαστικού χαρακτήρα για να προστατευτούν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να επικεντρωθούμε στις ε, ουσιώδες ε, νομοθετικές πράξεις, ε, να δώσουμε στην Κομισιέν κάποιο δυνατότητα ευελιξίας για τις μη ουσιώδες νομοθετικές πράξεις και όπως είπε ο κύριος Λάινεν βρισκόμαστε ακριβώς στο αυτό επίπεδο με το Συμβούλιο, δεν είμαστε κατώτεροι. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να τονίσω κάποιες πτυχές της ο Σάιγερ, τις οποίες θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Πρώτα απ' όλα, απορρίπτουμε τις διατάξεις που επιβάλλουν υποχρεώσεις συμπληρωματικές, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια του άρθρου 290. Τώρα, δεύτερη σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Τροπή για μια έγκαιρη και συνεχή υποβολή των εγγράφων. Τρίτον, η ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει έλεγχος αφού προηγούμενα θα έχουμε λάβει όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές το λόγο θα είχε κανονικά ο κύριος Ραπχάη, αλλά απουσιάζει, οπότε θα δώσουμε το λόγο στους Πρασίνους και στην κυρία Λίχτινμπεργκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Συχνά αυτά τα θέματα τα ε, θεσμικά, τα διαρθρωτικά, τα υποτιμούμε. Τα θέματα των σχέσεων στο διοργανικό τρίγωνο. Στην έκθεση αυτή, λοιπόν, τα θέματα αυτά τα ε, συνοψίζει εξαιρετικά ο κύριος ε, Σάγερ και ήταν πολύ καλή συνεργασία μας και επιθυμώ να τον ευχαριστήσω ειλικρινά γι' αυτό με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε πλέον νέες σχέσεις δημιουργήσει και αυτές οι νέες σχέσεις και ε, συσχετισμοί δεν θα πρέπει να ακυρωθούν από την πίσω πόρτα. Περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Η κεντρική ιδέα ποια ήταν ακριβώς η ισοτιμία μεταξύ Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να διατηρείται και να δημιουργείται και να εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις που εχωρούμε τις αρμοδιότητες και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά είναι εφικτά καταρχήν ε, διαδικαστικά και δεύτερον μπορούν ε, να είναι και εγγυημένα. Δηλαδή για μας η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που να το επιτρέπουν με τρόπο που να μπορούμε εγκαίρως να έχουμε τα έγγραφα στη διάθεσή μας για να λαμβάνουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Και να μην υπάρχει απλώς ε, μια συναντήληψη, μια συνεννόηση. Όχι, συμφωνία ε, συγκεκριμένοι για κάποια θέματα και να μην υπόκεινται στην πολιτική ε, αυθαιρεσία ή ε, συγκυρία ή στην εκάστοτε ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε κανόνες σαφείς, καλούς, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στην ουσία και στην πραγματικότητα και όχι να ε, λαμβάνουμε γνώση θεωρητικά. Ευχαριστώ κύριε Σάγια, ευχαριστώ λέει πρόεδρο και διακόπτει την ομιλήτρια. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σα. τώρα εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών. Ε, ο κύριο Ζόμπρο δεν είναι παρόν. επίση και εκ μέρου τη Ένωση, της ομάδας Ευρώπη για την Ελεύθερη Δημοκρατία, ο κύριος Ντάρτμουθ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Περισσότερο από ό,τι περίμενα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, αναφέρεται στο λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα ο εισηγητής. Ναι, η ελιτιστική όμως αυτή το ελιτιστικό αυτό οικοδόμημα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και με παραξενεύει πρέπει να σας πω το γεγονός ότι παρά την ευγλωτία του εισηγητή θεωρεί ότι είναι λύση το άρθρο 290 διότι εμείς το άρθρο αυτό το ερμηνεύουμε ως μια δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποκαταστήσει ή και να τροποποιήσει ακόμη ε, νομοθετικά έργα, νομοθετήματα. Πρόκειται για μια πολύ γενική δυνατότητα, ευρύτατη ε, δυνατότητα που μάλιστα είναι ανοιχτή και σε ευρύτατες ερμηνείες. Διασφαλιστικέ δικλείδε λοιπόν για, τον, για την κατάλληλη χρήση αυτών των εξουσιών που εκχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχουν κατά τρόπο επαρκή στα κείμενα τη συνθήκης. Ίσως θα μπορέσει να μας εξηγήσει μετά ο εισηγητή γιατί τις θεωρεί επαρκή αυτές τις διασφαλιστικές δικλείδε που εμεί δεν βλέπουμε. Περαιτέρω δε εκχώρηση εξουσία από το άμεσα εκλεγμένο στο Κοινοβούλιο στην μη σε επιτροπή δεν μπορεί να γίνει δεκτή ανεξαρτήτως του τι ισχυρίζεται ότι προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Εμείς διαρκώς υποστηρίζαμε και εξακολουθούμε να φρονούμε ότι δεν διαθέτει νόμιμο έρισμα η συνθήκη της Λισαβόνας καθώς δεν κυρώθηκε με διαδικασία δημοψηφίσματος που άλλωστε είχαν υποσχεθεί και τα τρία κόμματα εξουσίας στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο που όμως δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους και επίσης θα πρέπει να πω ότι το άρθρο 290 είναι προϊόν των συμβιβασμών της συνθήκης της Λισαβόνας δεν διαφυλάσσει τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και περιμένω να δω αν ο εισηγητής έχει επιχειρήματα για να αποκρούσει τις δικές μου θέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν από τους μία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, διακαής φιλοευρωπαϊστής θεωρώ ακριβώς ότι η συνθήκη της Λισαβόνας και για τα ίδια επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν μόλις τώρα είναι μια καλή συνθήκη γιατί διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να σταθεί και να πει τα λόγια αυτά και να προχωρήσουμε προς τις εξελίξεις που θα θέλαμε και για το μέλλον. Θα ήθελα να πω όμως ταυτόχρονα ότι θεωρώ ότι θα πρέπει και το άρθρο 290 να ε, μην οδηγηθεί σε μια ερμηνεία κατά την οποία το Συμβούλιο μπορεί να δώσει να εκχωρήσει νομοθετικό έργο αποκλείοντας από την απόφαση αυτή το, το Κοινοβούλιο. Είπε ο κύριος Σάιγερ βέβαια ότι είχαμε και χιλιάδες ακόμη νομοθετημάτων ε, κάθε εκχώρηση που περούσαν, ε, περνούσαν σε μια γκρίζα ζώνη απουσίας ουσιαστικά αρμοδιοτήτων για το ποιος θα ήταν αρμόδιος να τα κρίνει δηλαδή και εκεί που πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις ακριβώς για να απαντήσουμε στα αρνητικά επιχειρήματα των αντιευρωπαϊστών πρέπει να λαμβάνουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις, να προχωρούμε στο νομοθετικό μας έργο αποτελεσματικά. Αυτά τα βλέπω νομίζω ξεκάθαρα. Ξέρω αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε κι εσείς πολύ την ύπαρξη αυτού του Freedom of Information Act των Ηνωμένων Πολιτειών, της, ε, του νόμου για την ελευθερία στην ενημέρωση. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε copy-paste αυτό το νομοθέτημα και να το εισαγάγουμε στη δική μας νομοθεσία, πράγμα το οποίο θα μας επέτρεπε να ενημερωνόμαστε άμεσα για όλα αυτά τα νομοθετήματα τα οποία προχωρούν μέσα από τις διαδικασίες, τα χιλιάδες αυτών των νομοθετημάτων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε να προχωρήσουμε σε επαναστατικές μεταρρυθμίσεις στη δημοκρατική μας τάξη. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Βλέπω ότι δεν ζητεί κανεί από του συναδέλφου να λάβει το λόγο με τη δικασία του Καρστιάη. Η κυρία Τιτσάου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Με μικρόφωνο παρακαλώ κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να πω για το θέμα αυτό ότι είναι καινοτομία η συνθήκη της Λισαβόνας και το άρθρο 290. Τα νομοθετήματα που εκχωρούνται είναι γενικής φύσεως ε, που δεν μπορούν να αλλάξουν την ουσία ενός βασικού νομοθετήματος και ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ουσία δηλαδή ε, δίνουμε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσει ε, με μια ελάχιστη προθεσμία προσβολής ή κατάθεσης ένστασης και ορίζονται κάποιοι όροι και προϋποθέσεις. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να ασκήσουν ένα έλεγχο Μόνο όμως χωρισμένα νομοθετήματα, τα οποία μπορούν επίσης να δημοσιεύονται και να εκφράσουν αντιρρήσεις και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια όμως κύριε Επίτροπε. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και στην εκπόνηση αυτών των νομοθετημάτων. Άλλος κανείς συνάδελφος θέλει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ παρακαλώ. Όχι. Οπότε ε, θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον Επίτροπο κύριε Σεφσκοβίτς. Ελπίζω να σας είπα καλά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω τις παρατηρήσεις των μελών. Φυσικά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λάινεν ότι η συνθήκη Λισαβόνα ε, έφερε σημαντικές αλλαγές. Το τόνισε και ο εισηγητής κύριο ε, Σάγερ. Φυσικά και έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα ζητήματα που χωρούν στη διαδικασία και όλα αυτά θα συμβούν με απόλυτο σεβασμό προς τον νομοθέτη. Αυτό είναι πολύ καλό για την μελλοντική συνεργασία μας τώρα. Σε ό,τι αφορά τα κατεπήγον θέματα και τις κατεπήγουσες διαδικασίες, ε, θέλω να σας διασφαλίσω πως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σε έκτακτες ε, περιστάσεις ε, γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτών των ε, μέσων και δεν έχουμε τέτοια πρόθεση να το πράξουμε τώρα. Σε ό,τι φορά τα σχόλια του κυρίου Κοέλιο και της κυρίας Λίχτεμπεργκ να τους διαβεβαιώσω πως ε, θα κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας για να διασφαλίσουμε την αποστολή των εγγράφων ταυτόχρονα Προ το Κοινοβούλιο με τα έγγραφα τα οποία αποστέλουμε στο Συμβούλιο ότι όταν πρόκειται για οικονομικά ζητήματα πραγματικά το Συμβούλιο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε τώρα να αναπτύξουμε και μια νέα μορφή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προπαρασκευαστικέ εργασίε σε ό,τι αφορά τι κατεξουδότηση πράξη. Ω εκ τούτου λοιπόν θα δείτε αυτές τις ε, νέες ε, δυνατότητες στις ε, συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με το Συμβούλιο τώρα σε ό,τι φορά τις αρμοδιότητες αναφορικά με το 290 ότι αυτές δεν είναι ελέγξιμε. θα ήθελα να πω ότι εσεί αποφασίζετε κατά πόσον εξοδοτείτε πράξεις στην Κομισιόν ή όχι και εσείς μπορείτε φυσικά να καλέσετε αυτή τη δυνατότητα ή να ε, έχετε αντιρρήσεις ε, επί των προτάσεων που υποβάλλει η οχι και εσεί. μπορειτε φυσικα να καλεσετε αυτη τη δυνατοτητα η να εχετε αντιρρησεις επι των προτασεων που υποβαλλει η κομισιον Δεν νομίζω λοιπόν υπάρχει κάποια φαιά ζωή. Είναι, όλα καθορισμένα σαφέστατα στι ε, συνθήκε και η Κομισιόν πρόκειται να τα σεβαστεί. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Το λόγο έχει ο εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση και βέβαια τη συνεργασία όλες τις επιτροπές, ιδιαίτερα όμως την Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αναφέρω. Υπήρχε και πολλά νέα καθήκοντα για το μέλλον, αλλά και ιδιαίτερα συμβάλλει σε αυτέ τι ε, ε, εργασίε μα. Ιδιαίτερα δεν ευχαριστώ και τι ομάδε, πολιτικέ ομάδε για την καλή συνεργασία. Πρέπει να σα πω ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια διελκυστίνδα με το Συμβούλιο. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη διαφύλαξη και τη σαφή περιγραφή των δικών μα δικαιωμάτων και προνομιών. Βέβαια είναι πολύ πιο ε, ευχερής η επίτευξη αυτού του σκοπού εάν συμμερίζονται τις θέσεις και τις προσπάθειές μας και οι συνάδελφοι από τις άλλες ομάδες. Έτσι λοιπόν, ομόφωνα πρέπει να σας πω, μπορούμε να μιλήσουμε όλοι σήμερα και να διεκδικήσουμε τη διαφύλαξη των προνομιών μας. Ε, ο κύριος Επίτροπος μίλησε για, το, για την ευθυγράμμιση, το alignment. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει αυτή η συμπληρώση που χρειάζεται να λαμβάνουν χώρα όπου δεν υπήρχε μέχρι τώρα η συναπόφαση. Αυτό το ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι ήδη. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να έχουμε και την απρόσκοπτη πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, πράγμα το οποίο ήδη υπάρχει ως πρόβλεψη στη Διοργανική Συμφωνία, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε και τι είδους ε, διαβουλεύσεις και συνομιλίες λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο και να είμαστε ενήμεροι εγκαίρος. Για δε το είναι περιστολή των ε, αρμοδιοτήτων και προνομιών μας αγαπητοί συνάδελφοι δεν μπορώ να σας ε, πω τίποτα άλλο παρά να σας παραπέμψω στα ίδια τα κείμενα. Δεν μπορεί να ερμηνεύετε εσείς ότι περιστέλλονται οι εξουσίες μας με αυτά τα κείμενα, με αυτά τα άρθρα, με αυτό το άρθρο συγκεκριμένα συνθήκης Λισαβόνας. Ναι, είχαμε το πρόβλημα αυτό στο παρελθόν. Τώρα όμως το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει προσφυγή, μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να ανακαλέσει την εκχώρηση της νομοθετικής εξουσίας. Είμαστε η κυρίαρχοι αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Έχουμε την εξουσία να ασκήσουμε τις προνομίες και τα, τις αρμοδιότητές μας και είναι καθήκον μας να ασκήσουμε στην πράξη αυτές τις εξουσίες και αρμοδιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Τη συζήτηση την ολοκληρώσαμε έτσι και η ψηφοφορία θα λάβει στις Βρυξέλλες χώρα. Κυρίε και κύριοι, προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης σε μια προφορική ερώτηση συγκεκριμένα για προφορική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα της ασφάλειας των αερομεταφορών, μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εναέρειες μεταφορές.